προβλήματα. Γι' αυτό ε, καταλήγω και σε διαφορετικά συμπεράσματα από ό,τι άλλοι συνάδελφοι. Α, πρέπει να σταματήσει αυτή η βοήθεια. Αύριο στις 11.30. Περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση της κυρίας Νικόλ Κιλ για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία. Ήθελα να παρακαλέσω την ε, εισηγήτρια, την κυρία Κιλ να λάβει το λόγο να μας παρουσιάσει την έκθεσή της για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και τέσσερα χρόνια που εφαρμόζεται η στρατηγική για την Κεντρική Ασία έχουν γίνει πολλά πράγματα. Η Ευρώπη έχει θεσπίσει σταθερό και τακτικό διαλόγο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρωτοβουλίες και προγράμματα έχουν προωθηθεί για τους 7 τομείς που στοχεύουμε. Στα πλαίσια της ε, αραβικής ε, ε, επανάστασης, της κατάστασης στο Αφγανιστάν, για τα τραγικά επεισόδια στην Κυργυζία το 2010, τα όρια της στρατηγικής μας είναι πολύ πιο ορατά σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση. Το 2012 προβλέπεται η έκθεση της εξωτερικής υπηρεσίας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είπαμε να κάνουμε αυτή την έκθεση. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις αξίες της και τους στόχους της σε αποτελεσματικά προγράμματα. Δεν έχει ορατότητα, ε, δεν είναι... Ε, ε, έχει μια δειλή παρουσία δεν υποστηρίζουμε επαρκώς και ανοιχτά την κοινωνία των πολιτών, τα ανεξάρτητα ΜΜΕ και τους προασπιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές φορές κυβερνητικά ιδρύματα είναι αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται με τα κοινοτικά λεφτά και αυτό εις βάρος των πραγματικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι πεπισμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε μία νέα προσέγγιση της Ένωσης που θα βασίζεται στην ανθρώπινη ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία. Όλες μας οι δράσεις, σχέδια, πρωτοβουλίες θα πρέπει να έχουν ως μύτο την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Παίρνοντας παράδειγμα το τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν όπου ε, υποστηρίχτηκε το καθεστώς αντί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό του είδους η καταστολή όμως διαρκεί λίγο ή η Αραβική Επανάσταση το αποδεικνύει. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας και να απαντήσουμε στις ε, στις προκλήσεις ε, στην Κεντρική Ασία για να μην έχουμε τα ίδια πράγματα στο Καζακστάν εδώ και πέντε μήνες απεργούν οι εργάτες της πετρελοπηγές οι ε, πρόορες εκλογές που θα γίνουν τον Ιανουάριο γίνονται με ένα φόντο κοινωνικής ε, σύγκρουσης άνευ Έχουμε το κουράγιο και την τιμιότητα να πούμε στις αρχές του Καζακστάν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανασύρει τα κατάλληλα αποτελέσματα, συμπεράσματα συγγνώμη, όταν θα συζητήσουμε την εταιρική συμφωνία. Η Human Rights Watch ε, που ε, δημοσίευσε χτες μια έκθεση μας σκανδάλισε σχετικά με τα βασανιστήρια, τα πίστευτα βασανιστήρια στην Τασκένδη, στο Ουζουμπεκιστάν όπου έχουν συλληφθεί ε, προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ έρχεται η κυρία Άστον και μας λέει κάθε φορά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν τον λόνα των εξωτερικών μας δράσεων. Ζητούμε λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση των πολιτικών μας προς την Κεντρική Ασία. Εγώ είμαι ιδιαίτερα περήφανη για το γεγονός ότι αυτό το κοινοβούλιο έθεσε την αιρεσιμότητα και την αρχή διαφοροποίησης στην καρδιά της νέας μας προσέγγισης συστήνοντας να εντείνουμε την υποστήριξή μας ε, στην κοινωνία των πολιτών και στα ανεξάρτητα ΜΜΕ. Θα μπορούσε λοιπόν, ε, δεν μπορεί μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρεται τίμια σε μια περιοχή και να γνωρίζει σε μια άλλη περιοχή τις ίδιες αξίες όταν αυτές παραβιάζονται. Χρειάζεται μια διαβουλευμένη προσέγγιση για τις εθνικές σειράξεις. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το εμπόριο όπλων, με τη διακίνηση ναρκωτικών, με το σωματεμπόριο, με, την, με το νερό. Όλα αυτά απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Κεντρική Ασία αλλά και στην Ευρώπη. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή, να διευκολύνει στον διάλογο και να δημιουργήσει ένα φόρουμ, ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ ad hoc που η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την αντιπροσωπεία της ε, μέσα από την μεικτή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία θα μπορούσε να προτείνει στους εταίρους της Κεντρικής Ασίας ώστε να συναντιούνται όλοι μαζί. Έχω πέντε συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο και πρώτα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κέλλη. Εμένα μου αρέσει αυτή η έκθεση. Προσφέρει πολλά και για την ευρωπαϊκή στρατηγική και ιδιαίτερα για τις πέντε χώρες που αφορά. Από τότε που πρωτοακούστηκε αυτή η έννοια της στρατηγικής αυτής της Ένωσης υπήρξαν, έγινε μεγάλη πρόοδο στην Κεντρική Ασία. βελτιώθηκε η ένομη τάξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Είναι περιοχή που έχει στρατηγική σημασία και για μας και είναι, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να συνάψουμε στενότερους δεσμούς. Ιδιαίτερα θα ήθελα να γίνονται τακτικότερα διασκέψεις Ένωσης Κεντρικής Ασίας. Πρέπει βέβαια να δούμε τι πρόοδο θα σημειώσουμε και στο μέλλον. Θέλει κυρία Τικάου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Datorită potențialului comercial și de securitate energetică al Asiei Centrale, precum și a interesului comun al țărilor din Η ενεργειακή ασφάλεια τη Κεντρική Ασία είναι κοινό συμφέρον και των χωρών τη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι εξαγωγέ και τη συνεργασία, τη βιώσιμη οικολογική ανάπτυξη με βάση τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ένωσης. Η Κασπία, το Αζερβαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν είναι σημαντικές αιστείες φυσικού αερίου και το σχέδιο Ναβουχοδονόσορ που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχέδιο που θα συμβάλλει στην καλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα της Ένωσης. Μια καλύτερη λοιπόν διακυβέρνηση των πόρων αυτών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή ανάπτυξη στην περιοχή και γι' αυτόν τον λόγο υποστηρίζω τις συμφωνίες αγοράς τέτοιων του φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα με μεγάλη βέβαια διαφάνεια της λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων. Καλό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς μας οδηγούν να υποθέσουμε ότι παραβιάζονται συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης στο Καζακστάν. Και έχω μαρτυρίες. Στις 26 Οκτωβρίου του 2011 ένας δημοσιογράφος και ένας κάμεραμαν ε, στο Μάτζισταου ε, έπεσαν ε, θύματα μιας τρομοκρατικής δράσης. Αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι είχαν ξεκινήσει ένα πρακτορείο το οποίο για χρόνια πληροφορούσε με ασφαλείς ειδήσει για τα διαμοιβόμενα στην Κεντρική Ασία οι δολοφόνοι τους ε, κλέψανε και το φορητό υπολογιστή των δημοσιογράφων που είχαν μέσα ένα σωρό στοιχεία για το τι γίνεται με τη διαχείριση των πετρολοπηγών. Ζητώ από την Κομισιόν να καταδικάσει αυτού του είδους τις πρακτικές και να τις λάβει υπόψη στις διαπραγματεύσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποστηρίξει την ελευθεροτυπία σε αυτές τις χώρες και να γίνει ε, με, ε, μια στρογγυλή τραπέζα τραπέζα με τους εκπροσώπους του Καζακστάν, των εργαζομένων στην περιοχή του Ματζεστάου και με τις πετρελαϊκές εταιρείες για την απεργία. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή. Είμαι μέλος της αντιπροσωπείας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και με μεγάλη χαρά δέχομαι τις βασικές αρχές αυτής της στρατηγικής. Αλλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να απαντήσουμε το ερώτημα ε, του πώς θα προωθηθούν αυτά πιο αποτελεσματικά αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σημαντικοί παράγοντες στη διεθνή σκηνή. Οι δραστηριότητες μας μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές όσο και των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΕΔΕ ενεργειακός τομέας, ο αγωγός Ναβουχοδονόσορ, ε, καθυστερεί δυστυχώ, οι Κινέζοι έχουν διαφορετικό αγωγό προβλέψει και προχωρούν πιο γρήγορα από μας. Πρέπει λοιπόν κάτι παραπάνω να κάνουμε. Μπορούμε νομίζω να συμβάλλουμε πολύ θετικά στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και στην ανάπτυξη των χωρών αυτών καθώς και στη δημοκρατική τους διακυβέρνηση η εμπειρία μας μπορεί να είναι πολύτιμη και για την οικονομία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στην περιφέρεια αυτή, στην περιοχή αυτή υπάρχει ισχυρή επιρροή της Ρωσίας και η παράδοση μιας ρωσικού τύπου διακυβέρνησης. Αν θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την περιοχή αυτή πρέπει να είμαστε παρόντες εκεί και να ασκούμε και εμείς την επιρροή μας σταθερά. Αλλιώς θα αφήσουμε την περιφέρεια σε χώρες σαν τη Ρωσία και την Κίνα και οι κάτοικοι εκεί δεν θα έχουν άλλη εναλλακτική λύση ούτε κανένα όραμα καλύτερης κοινωνίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε εκεί στην παρουσία μας και να προσπαθήσουμε να συμπιάσουμε την οικονομική συνεργασία με τη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών αν πιστούν ότι τα προγράμματά μας είναι πιο ωφέλιμα για εκείνες θα είναι πιο προετοιμασμένες να εφαρμόσουν και πιστότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν τα προγράμματά μας τους ωφελήσουν θα δεχτούν και τα κριτήριά μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δομής της κοινωνίας τους. Με συνδυασμένο λοιπόν τρόπο και να μην περιμένουμε από τη μια μέρα στην άλλη βελτιώσεις. President, uh, Uh, Κύριε Πρόεδρε, σε την μέλη, ε, χαιρετίζω το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κεντρική Ασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί η Κεντρική Ασία είναι μια περιοχή που όσο πάει αυξάνει τη σημασία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, την τρομοκρατία, τα ναρκωτικά και άλλα εγκλήματα. Μια οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση είναι πρόκληση όχι μόνο για τις λόγω χώρες, αλλά και για την περιφερειακή συνεργασία και ασφάλεια. Ταυτόχρονα όμως η περιφέρεια εκείνη είναι πλούσια σε πρώτες ύλες. και μπορεί να συμβάλλει στην ε, ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ενδιαφέρον ε, μεταξύ των ε, κρατών εκεί να ενδυναμώσουν την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τη συνεργασία του 2007, η Κομισιόν με λίγους πόρους και σε λίγο χρονικό διάστημα μπόρεσε να βελτιώσει το ρόλο της συνεργασίας με την Κεντρική Ασία. Μέσα στα πλαίσια του ΕΕ βοήθησε στην Κυριακή Δημοκρατία να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα της σημασίας της ε, αυξημένης δέσμευσης. Η στρατηγική αυτή οδήγησε και σε άλλες αξιόλογες ε, εξελίξεις. Διάλογο υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Ασίας περιφερειακά σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Επίσης, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις πέντε χώρες. Για την ενέργεια έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ την πραγματοποίηση της υπερκαυγασίας ε, του υπερκαυσινού αγωγού. Ε, όσον αφορά το είδωρ, βελτιώνουμε την ε, κατάσταση της συνεργασίας μέσω διαλόγου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση εμπλέκεται πάρα πολύ στην ε, μεταρρύθμιση της παιδείας σε πολλές από τις χώρες αυτές. Τα προγράμματα τεχνικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών είναι ένα από τα κύρια διεθνή προβλήματα της περιοχής. τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο και οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να είναι κύριοι επενδυτές ε, στην περιοχή εκεί και διευρύναμε την εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να επενδύσει εκεί στον τομέα ιδίως της ε, ενέργειας και του περιβάλλοντος στο Κυργιστάν, Τατσίρισταν και Ουσμπεγιστάν, προωθούμε στρατηγικές μέτρες και στο Ουσμπεγιστάν για το μέλλον. Η περιφέρεια αυτή ευρέω εξακολουθεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Πολλά θα πρέπει ακόμα να γίνουν όσον αφορά τη σχέση μας με την, με την περιοχή. Η κατάσταση ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανησυχητική, όπως είπε και η κυρία Φάνα. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα τη δέσμευσή μας σε αυτό τον λεπτό και σημαντικό τομέα. Προσπαθούμε να αυξήσουμε την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσουμε κοινοτικά προγράμματα πολύ περισσότερα λόγω του σχετικά περιορισμένου των πόρων μας στην περιοχή αυτή. Ο συντονισμό ε, της ε, συνεργασία με άλλου διεθνού δωρητέ θα πρέπει να ενδυναμώται συνεχώ. Το γεγονό ότι οι πόροι μα είναι περιορισμένοι καθιστούν όσο πάει και πιο σημαντικό το να εστιάσουμε την ενίσχυση που δίνουμε, όπως τονίζεται και στην ε, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας από τους κύριους ε, στόχους είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Και η, κύριος, η Δημοκρατία, ο κύριος και το κύριο Σταν είναι εκείνοι που ωφελούνται περισσότερο γιατί είναι οι πιο φτωχές χώρε. Είναι πολύ διαφορετική η περιοχή εκεί και παρόλο που προωθούμε τη συνεργασία στο περιφερικό επίπεδο, παραδείγματο όσον αφορά ε, το θέμα της διαχείρισης των συνόρων του ύδατος και την καταπολέμηση του αθλητισμού ναρκωτικών, προσπαθούμε να ε, βοηθήσουμε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Με το Καζαστάν, παραδείγματο χάρη. Ανοίξαμε πρόσφατα διαπραγματεύσεις για ενδυναμωμένη συμφωνία ε, εταιρική σχέση και συνεργασία που θα είναι η πρώτη στην περιοχή αυτή. Και ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να σα πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να παίξει όταν προχωράμε στη σχέση μα με την Κεντρική Ασία. Χαιρετίζουμε τι επισκέψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περιοχή αυτή και τον τεχνικό διάλογο καθώς επίσης και την δέσμευση του Κοινοβουλίου προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας δίνει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την αναθεώρηση των σχέσεων μας και συγχαίρω τον εισηγήτρια. Η συζήτηση έληξε και η ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Κιλνίλσεν θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση της κυρίας Καριμάντελη για την υγεία και την ασφάλεια